με θέμα την ετήσια έκθεση του 2013 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το τομέα. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Παντσέρη, για τέσσερα λεπτά. Πρέγκο κύριε Παντσέρη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η έκθεση αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο αξιολόγηση ε, των πολιτικών που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα να απογραμμίσω την πολύ σημαντική δουλειά που έχει κάνει ο ειδικό απεσταλμένο. Με αυτή λοιπόν την ε, έκθεση ε, έχουμε μια θεματική και γεωγραφική προσέγγιση και θεωρώ ότι αυτή η έκθεση είναι πολύ χρήσιμη γιατί εντοπίζει κάποιε κατευθυντήρε γραμμέ για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τους μεμονωμένους επιτρόπους. Αγαπητοί συνάδελφοι, το 62 στη Βιέννη Είχαμε έναν ε, νομικό φιλευθερισμό, τον αγώνα για τα δικαιώματα και αργότερα αυτό, ε, όπως ξέρετε, ακολούθησε και με άλλες πράξεις προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τον φασισμό. Εγώ όμως θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να μιλάμε για τον αγώνα των δικαιωμάτων. Προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων μέχρι και την ε, διαμαρτυρία των νέων στο Χονγκ Η Άννα Χάρεντ είπε το δικαίωμα να έχει κανείς δικαιώματα. Για να αποφύγουμε λοιπόν όλα αυτά αυτά να είναι απλά ένα σλόγγαν. Θα πρέπει να θυμηθούμε την πλήρη φράση που είναι το δικαίωμα να έχει κανείς δικαιώματα ή το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να εντάσσεται στην ανθρωπότητα. Και αυτό πρέπει να το εγγυάται η ίδια η ανθρωπότητα. Είναι λοιπόν σαφές ότι η ύπαρξη δικαιωμάτων είναι επιτακτική ε, και Θεωρώ ότι αυτή η πολιτική για την οποία μίλησαν σχετικά με τις διακριτικές μεταχειρήσεις βάρος των ομοφυλοφίλων ε, αυτό υπάρχει και σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις. Στη σημερινή εποχή τα δικαιώματα είναι κάτι απολύτως απαραίτητο αλλά θεωρείται και πολυτέλεια στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης η οποία αντιμετωπίζεται μόνο με δημοσιονομικά μέτρα. Έχω κατά νου κυρίως ε, τις χώρες της γειτονίας μου και διαρωτώ με τη στιγμή όμως όπου ε, δεν υπάρχουν δικαιώματα ή απομακρύνονται τα δικαιώματα. Τελικά τι ακριβώς επιδιώκουμε όταν περιορίζονται τα δικαιώματα που αφορούν την εργασία, την υγεία, ε, την ε, παιδεία, τα αστικά δικαιώματα, αυτό κατ' ουσίαν είναι επέμβαση κατά της δημοκρατίας. Δεν είναι μόνο τα δικαιώματα που είναι αναπαλωτρίωτα, είναι και δικαιώματα που έχουν άμεση σχέση με την οικονομία. Αυτές λοιπόν οι σκέψεις για τα δικαιώματα μας οδηγεί σε μια πολιτιστική συζήτηση, μια συζήτηση η οποία αποκαλύπτει ότι υπάρχουν ε, νέες αναφορές σε αυτή την κρίση, οι οποίες αναφορές έχουν καταστήσει ακόμα σαφέστερη την σύγκρουση που υπάρχει, τη σύγκρουση όπου πρέπει κανείς να έχει κατά νου την εξέλιξη της ε, κοινωνίας. Με αυτή λοιπόν την έκθεση θέλουμε να στείλουμε ένα απλό μήνυμα ότι τα δικαιώματα δεν περιορίζουν τη δημοκρατία αλλά επιβάλλουν το ότι πρέπει να σκεφτούμε πώς ακριβώς πρέπει να να κινείται η πολιτική ευθερεσία. Σε τέτοιους ε, χαλεπούς καιρούς τα κριτήρια θα πρέπει να βασίζονται στην υποχρέωση να είναι δυνατή η εφαρμογή και ο σεβασμός των δικαιωμάτων. Γιατί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε δεν είναι ότι υπάρχουν υπερβολικά δικαιώματα, αλλά η άρνησή τους, δικαιώματα που δεν υφίστανται πλέον λόγω της βίας κατά των γυναικών, λόγω της φτώχειας, όλα αυτά ακυρώνουν την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Άρα δηλαδή υπολείπονται πάρα πολλά. Εγώ θεωρώ ότι το καθήκον της Ευρώπης είναι να κρατάει υψηλά την πρόκληση, να δείχνει συνέπεια για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτή την απειλή εις βάρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα μέρη του κόσμου. Σας ευχαριστώ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην υπάτη εκπρόσωπο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και όλους ε, όσους συνεργάστηκαν μαζί του. Ε, θεωρώ ότι ήταν ε, πάρα πολύ χρήσιμο το να ε, παρακολουθείτε τη δουλειά μου στο ε, θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν ήθελα να πω ότι συμμερίζομαι όχι μόνο την ανάλυση που κάνατε αλλά και αυτή την πρόσκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που ήταν να παραμείνει υψηλά η πρόκληση να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα, μικρά βήματα έστω σε περιπτώσεις όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα είτε παραβιάζονται είτε αμφισβητούνται και θα συνεχίσω στα αγγλικά. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να λαμβάνω μέρος σε αυτήν την ετήσια συζήτηση για την ετήσια έκθεση με θέματα δικαιώματα στο, τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο. Και όπως αναφέρει η έκθεση, η Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρει ότι θα πρέπει να, να αναγάγουμε την ε, αξιοπρέπεια στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας. Αυτή είναι η βασική μας προτεραιότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εξωτερικές μας δράσεις. Και θα έλεγα ότι αυτή είναι η πρωταρχική μας προτεραιότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και όχι μία από τις προτεραιότητες. Θα πρέπει να είναι το θεμέλιο ε, όλων των σχέσεων μας με τις τρίτες χώρες. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αισθενίζεται αυτό το στόχο, γιατί ανέκαθεν ε, προωθούσε τα ανθρώπινα δικαιώματα και στο καθημερινό έργο και με συγκεκριμένε δράσει. Καταρχήν, επισκεπτόμενοι χώρε που απειλούνται αυτά τα δικαιώματα. Ε, Επίσης είναι πολύ συμβολική η αξία του βραβείου Ζαχάροφα. Όλες αυτές οι δράσεις είναι βασικές, βασικές συνιστώσεις της κοινοβουλευτικής διπλωματίας που είναι απαραίτητη στη γενική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο εξακολουθούν να είναι πρόκληση. Και συμφωνώ ότι έχουμε σημειώσει πρόοδο σε πολλά σημαντικά θέματα, ιδιαίτερα μετά την έγκριση του πακέτου για τα ανθρώπινα δικαιώματα το 2010 και μετά το πρώτο σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την περίοδο 2012-2014. Θα πρέπει να υλοποιήσουμε πολλούς σημαντικούς στόχους. Και όλοι οι ευρωπαϊκοί φορείς ε, είναι στρατευμένοι υπέρ της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε εφοδιαστεί με τα εργαλεία για να εφαρμόσουμε ε, και να συνεκτιμούμε τη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις εξωτερικές μας πολιτικές. Και έχουμε εξαγγείλει την ε, προβολή μας ε, και την αξιοπιστία μας στον τομέα αυτό, επισημένοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα ως προτεραιότητες σχέση με τους εταίρους. Η δική σας υποστήριξη στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης ήταν κέρια. Τώρα θα πρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω και επίσης να διαρθρώσουμε το κοινό μας έργο με βάση ε, συγκεκριμένες προτεραιότητες. Από την ανάληψη των καθηκόντων μου προώθησα το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ξεκινώντας από τη διαμόρφωση ενός σχεδίου δράσης, που θέλω να στηρίζεται όχι μόνο σε ένα κατάλογο δράσεων, αλλά σε πολιτικές προτεραιότητες. Και στο πλαίσιο αυτό, μία από τις προτεραιότητές μας θα πρέπει να είναι η υποστήριξη ε, των διαδικασιών δημοκρατικής μετάβασης και οι δικές σας προσπάθειες και το έργο σας θα πρέπει να στηρίζει το δικό μας. Και χαίρομαι που στην έκθεσή σας ε, εκτιμάτε τις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τακτική ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε διάφορες ε, περιπτώσεις. Και επίσης θέλουμε οι οργανώσει κοινωνία των πολιτών αποτελούν βασικό μα εταίρο με τις οποίες έχουμε διαβουλεύσει. Οι διαβουλεύσει με την κοινωνία των πολιτών πριν και μετά διαλόγου ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι σημαντικές πολιτικές ε, ε, συνιστώσεις της πολιτικής. Και μετά ε, και έχει αποτελέσει συστηματική πρακτική και στο, ανθρώπινο, και στο Συμβουλίο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και πέρυσι είχαμε αντίστοιχη συμμετοχή πάνω από 200 οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών και με ιδιαίτερο θέμα την ελευθερία έκφρασης. Χαίρομαι ιδιαίτερος που συμφωνούμε ότι είναι αξιέπαινη δράση του Ευρωπαϊκού του Ευρωπαίου Εντεταλμένου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, του πρώην συναδέλφου σα, του Σταύρου Λαμπρινίδη. Παρόλο που κάθεται δίπλα μου, ε, θα ήθελα να επενέσω το έργο του, γιατί είναι ανεκτήμητη η προσπάθειά του στην πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Γιατί έτσι διευρύνουμε περιφερειακού μηχανισμού και προωθούμε την οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και με ιδιαίτερη χαρά σα αναγγέλω εδώ και επίσημα ότι αποφάσισα να παρατείνω την εντολή του ειδικού εντεταλμένου και μάλιστα το Συμβούλιο ενέκρινε αυτή την απόφαση. Και επανέρχομαι στο κοινό μας έργο, της θέσπισης προτεραιοτήτων για τις δράσεις μας στα ανθρώπινα δικαιώματα. Να επισημάνω τα εξής. Καταρχήν, συμφωνώ και στερίζομαι πλήρως την προσέγγισή σας. Θα πρέπει να επικεντρώσουμε τι προσπάθειές μας για να βελτιώσουμε την εσωτερική και εξωτερική μας συνοχή. Αν θέλουμε να ενισχύσουμε την αξιοπιστία της Ένωσης ως παγκόσμιο φορέα, θα πρέπει να εξετάσουμε τον αντίκτυπο που έχουν οι πολιτικές μας τα ανθρώπινα δικαιώματα και εκτός των σύνορων μας. Και επίση ε, οι προσπάθειε μα, ε, οι εξωτερικέ, θα πρέπει να είναι συμπληρωματικέ. Ε, με το έργο του Αντιπρόεδρου Τίμερμανς, ώστε όλες οι κοινοτικές πολιτικές να συνάδουν με τη χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να είμαστε συνεπείς ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και εντός και εκτός των συνόρων μας. Και πάνω απ' όλα εντός των συνόρων μας για να είμαστε πραγματικά αξιόπιστοι και στις εξωτερικές μας δράσεις. Ως προς τις προτεραιότητες, διαβάζοντας την έκθεσή σας, αναγνωρίζω κι εγώ και οι δικές μου προτεραιότητες ε, του σχεδίου δράσης. Μερικά παραδείγματα πέραν της ανάγκης ε, ενίσχυσης ε, της εσωτερικής και εξωτερικής συνοχής των πολιτικών μας, θα ήθελα να σας αναγγείλω την υποστήριξή μας στην κοινωνία των πολιτών, την πολιτική, τεχνική και οικονομική ε, συνδρομή και ενίσχυση των προσπαθειών για να διευρυθεί ο χώρος για τις οργανώσεις αυτές που συρρυκνώνεται σε πολλές χώρες. Επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις κατάφορες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που γίνονται σε ένοπλες συγκρούσεις και κρίσεις γύρω μας. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ε, προλάβουμε τέτοιες παραβιάσεις και να ε, βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα διεθνών μηχανισμών για να αντιμετωπίσουμε την ατιμορρησία. Η πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι ένα αφηρημένο εγχείρημα. Έχουμε συγκεκριμένου μηχανισμού που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά θα πρέπει να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά του. Και λίγα λόγια σχετικά. Μέσω των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα ήθελα ε, να μην περιοριστούμε όμως ε, μόνο εκεί. Θα ήθελα σε όλες τις ε, διμερείς επαφές μας με τις χώρες εταίρους να περιλαμβάνουμε και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και το έργο του κυρίου Σταύρου Λαμπρινίδη συνάδει και με την δική μας δέσμευση για τις αντίστοιχες σχέσεις με συνομιλητές και χώρες εταίρους. Επίσης, θέλω να αναβαθμίσω την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών, των γυναικών, των ΛΟΑΔΜ, αλλά και της ελευθερίας έκφρασης, της ανεξιθρησκείας, μέσω κατευθυντήριων γραμμών ώστε να ε, έχουμε ε, αφύπνιση όλων των αρμοδίων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ευαισθητοποίηση. Επίσης, ειδικέ αντιπροσωπείες ε, που έχουν στενές επαφές με πολλές χώρες ανά τον κόσμο θα πρέπει και αυτές να επικεντρωθούν περισσότερο στη πρόθεση αυτών των αξιών και δικαιωμάτων και μπορούμε να συντονίσουμε αντιστοίχως τις προσπάθειές μας. Πέμπτη προτεραιότητα στο πλαίσιο τη προώθηση τη οικουμενικότητα και του αδιαίρετου χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα προωθήσουμε ταυτόχρονα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά δικαιώματα και μέσω της αναπτυξιακής μας βοήθειας. Και στο πλαίσιο αυτό πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποτελέσει πρωταγωνιστή και να πρωτοστατήσει σε αυτές τις προσπάθειες συνδυάζοντας τη, την εμπορική διάσταση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη σχετική πρόταση με την κοινωνική εταιρική ευθύνη. Σε ό,τι αφορά τι θρησκευτικέ μειονότητε, μίζων μέρημνα και μαζί με τους εταίρους ξεκινήσαμε μια προσπάθεια να καταπολεμηθεί η βία που διαπράτεται στο όνομα της θρησκείας και φυσικά να αντιμετωπιστούν τα αίτια, είτε αυτά είναι κοινωνικά, είτε οικονομικά, είτε πολιτικά. Για να δούμε πού οφείλεται η ριζοσπαστικοποίηση στις κοινωνίε μας και στη Μέση Ανατολή, αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου, όπως το Πακιστάν και το Αφγανιστάν. Επίσης, ε, θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχει πρόβλημα και στις δικές μας κοινωνίες. Και εκεί θα πρέπει να ενισχύσουμε την εσωτερική και εξωτερική διάσταση των πολιτικών μας. Η προώθηση της ελευθερίας ε, έκφρασης και της ανεξιθρησκείας θα πρέπει να είναι το βασικό στοιχείο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και αναπόσπαστο τμήμα της. Δεν νοείται ασφάλεια και σταθερότητα χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα. Και θα πρέπει να έχουμε υπόψη αυτό το γεγονός και να το υπενθυμίζουμε και στους εταίρου μας καθημερινά. Τους τελευταίους μήνες καταδικάσαμε ρητά τις κατάφορες και μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις οποίες προβαίνει το Ισλαμικό κράτος. Και προσπαθήσαμε να συνάψουμε συνασπισμούς και συμμαχίες για να καταπολεμήσουμε αυτή την τρομοκρατία. Μάλιστα έχουμε ε, πρωτοστατήσει και στη διεθνή ε, απάντηση στην ανθρωπιστική κρίση της Συρίας και επίσης ε, έχουμε εμπλακεί και στο Ιράκ. Και στη φετινή μας ανθρωπιστική ενίσχυση θέλουμε να φτάσουμε σε περιοχές όπου υπάρχουν μεγάλες ανάγκες και ευάλωτες ομάδες. Στη Συρία, σε περιοχές που δεν υπάρχει τόσο έντονη βία, προσπαθούμε να τρομολογήσουμε συγκεκριμένα προγράμματα για μειονότητε για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων και να διευκολύνουμε Μία μετάβαση που δεν θα αποκλείει κανέναν, λαμβάνοντα υπόψη τι ανάγκε και την επανένταξη των ευάλωτων ομάδων στην κοινωνία. Επίση, στηρίζουμε προσπάθειε ατοπικών φορέων, ώστε οι παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων να τεκμηριώνονται για να υπάρξει συνέχεια λογοδοσία. Είμαι ευγνώμων για τις ε, πολύτιμες προτάσεις και συστάσεις που περιέχει η έκθεσή σας και προσβλέπω στην υποστήριξή σας για να βρούμε τρόπους και να τις εφαρμόσουμε από κοινού και περιμένω με αδημονία τη συνέχιση της συζήτησης για να εμπλουτίσουμε ακόμη περισσότερο τις ιδέες μας. Ο, ο λόγος στην κυρία Χαουταλά. Για ένα λεπτό. Εκ μέρους Επιτροπής ΔΕΒΕ. Πάντοτε είναι σημαντική ημέρα μέρα που συζητάμε την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα εδώ στο Κοινοβούλιο. Και είναι η χαρά μου να πω εκ μέρους Επιτροπής Ανάπτυξης ότι ο κύριος ε, Παντσέρη ε, ενέταξε όλες τις ε, ανησυχίες μας ε, και τα σχόλιά μας στην ετήσια έκθεση. Είμαι σίγουρη ότι και είπα ότι εκπρόσωπος αντιμετωπίζει την αναπτυξιακή πολιτική ως αναπόσπαστο νήμα της εξωτερικής μας πολιτικής. Είμαι περήφανη που ε, διορίστηκε ο κύριος Σταύρος Λαμπρινίδης ως ε, ε, ειδικό εντεταλμένος. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ σωστή αυτή η απόφαση που ελήφθη από την προκάτοχο της είπατης προσώπου. Συγχαρητήρια. Ο κ. Παντσέρη στην έκθεση του δείχνει πως υφίστανται πολλά θέματα πριν δικαιωμάτων που σχετίζονται με την αναπτυξιακή πολιτική. Επίσης είμαι βεβαιά ότι εσείς ε, κύριε Πατή εκπρόσωπε, ε, ε, είσαστε σε άμεση επαφή με την αντίστοιχη γενική διεύθυνση της Κομισιόν. Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν τμήμα της ανάπτυξης. Αυτό είναι τόσο προφανές που δεν αναφέρεται καν στην έκθεση. Ε, και οι προτεραιότητες ε, τις οποίες, τις οποίες αναφερθήκατε αντιστοιχούν σε αυτά που το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Ανάπτυξης θεωρούν σημαντικά. Ευχαριστώ. Κυρία Ζητμάνσκα, για ένα λεπτό. Εκ μέρους της Επιτροπής Νομικών, υποθε... Νομικών Θεμάτων. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύουμε ότι τα βασικά δικαιώματα αφορούν τις ε, γυναίκες. Το 95% θα πούνε ότι όσον αφορά το θέμα αυτά τα δικαιώματα ε, Μεγάλο πρόβλημα είναι η παραβίαση δικαιωμάτων των γυναικών και θέλω να σας εξηγήσω τι ακριβώς ε, θεωρώ στο θέμα της βίας κατά των γυναικών. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει στα διάφορα κράτη να υπάρχει εμπιστοσύνη. Οι γυναίκες δεν θα πρέπει, πρέπει να είναι θύματα βίας. Οι γυναίκες δεν θα πρέπει να δίνουν την εντύπωση ότι δεν συνέβη τίποτα. Επίσης, τα κράτη-μέλη πρέπει να εκπαιδεύσουν προσωπικό, αστυνομίες και άλλους αρμόδιους για να μπορούν να βοηθήσουν ταχύτατα τα θύματα. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό για μας είναι ότι θα πρέπει να αλλάξουμε το σκεπτικό των νέων ανθρώπων. Αυτό όμω δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με νομοθετικά μέτρα. Εναπόκειται σε εμά να αλλάξουμε στάση. Πολλοί από εμά ερχόμαστε από όπου τα Τουκιά είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να, κάνουμε, να δώσουμε θάρρος στις ε, γυναίκες. Ευχαριστώ. Ο λόγος στον, στους των πολιτικών ομάδων τώρα. Ξεκινάμε ε, καταρχήν να σας ζητήσω να περιορίζεστε στο χρόνο το οποίο, σα, τον οποίο σας δοτίδουμε. Λόγος του κύριου Πέντε για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν να συγχαρώ τον ε, ε, εισηγητή τον κύριο Παντζέρη. Ε, για αρκετούς μήνες ε, συζητήσαμε αυτή την έκθεση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οπότε μπορώ να πω με χαρά ότι το κείμενο το οποίο θα κληθούμε να ψηφίσουμε αύριο αντικατοπτρίζει ορθά την ανησυχία του ΕΛΚ για την προστασία και την προωθήση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας και επιμένω ότι στο διτό χαρακτήρα. Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία. Πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά αποτελούν τμήμα ενός συνόλου. Και αυτό είναι το σημείο αφετηρίας της έκθεσης αυτής. Η έκθεση Παντζέρη ε, τονίζει πολύ σωστά την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Θα έπρεπε να είμαστε περήφανοι ε, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε αυτά τα δύο ζητήματα. Και το λέω και κατόπιν και στραχώδους συζητήσεως που έλαβε η χώρα προηγουμένως ε, όπου δυστυχώς κάποιος από τους συναδέλφους ισχυρίστηκε ότι από πλευράς δημοκρατίας η Ρωσία είναι σε καλύτερη θέση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση αυτή καταδεικνύει ότι αυτό είναι λανθασμένο ως ισχυρισμός. Τόσο σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία όσο και σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να προσθέσω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο και ταυτόχρονα ε, είναι υποχρεωμένη να σέβεται αυτά τα δικαιώματα εντός της επικράτειάς της. Όμω η έκθεση αυτή δεν αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντό Ευρωπαϊκή Ένωση και εντό των κρατών μελών. Το λέω αυτό διότι συζητούσαμε με του ε, συναδέλφου τη Επιτροπή ε, Πολιτικών Ελευθεριών που προφανώ ε, εξαιτία του ρόλου του ανησυχούν για το θέμα των δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα δεν θα πρέπει να υποδεικνύει τι θα κάνουν όλοι οι υπόλοιποι για την ομοποίηση των αμβλώσεων ή των γάμων μεταξύ των ομοφυλοφίλων για ηθικά θέματα. Δηλαδή θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Και ο κ. Παντζέρη ήταν πολύ θετικό σε ό,τι αφορά αυτή την ανησυχία. Κυρία Βαλενσιάνο, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συζητούμε μια εξαιρετική έκθεση. Από την δική μου πλευρά είναι μια έκθεση η οποία είναι αντικειμενική, είναι, ε, κάνει σε μια σε βάθος ανάλυση. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε και πολλά ευχάριστα νέα από τα πλευρά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, ξαναγεννώνται κάποια τέρατα τα οποία νομίζαμε ότι είχαν ε, νικηθεί. Ε, η έλψη ανεκτικότητας, ο ρατσισμός, ο φανατισμός και τα ανθρώπινα δικαιώματα απειλούνται. Αυτό δεν είναι μόνο λόγια αλλά και πράξη, είναι μια διαπίστωση. Γι' αυτό τον λόγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δηλώσει ρητά και απερίφραυστα ε, την δέσμευση, την προσήλωσή του στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου για την προστασία τους. Ε, για τις αρχές της δημοκρατίας και της αξιοπρέπειας για, όλα τα, για όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η οικονομική κρίση βοηθούν ε, σε ορισμένε περιοχές του κόσμου να συρρυκνώνονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα πρέπει να αναλάβουμε μια δέσμευση, δέσμευση για τη χρήση του κράτου δικαίου προκειμένου να προασπίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα πέραν της προτεραιότητάς μας που ασφαλώ είναι η ασφάλεια όλων. Ε, η δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η συλλογική συνέπεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεν είναι δυνατόν, όπως συμβαίνει μερικές φορές, από τη μια μεριά ε, να καταδικάζουμε και από την άλλη μεριά με το άλλο χέρι να υπογράφουμε συμφωνίες. Ε, όχι λοιπόν σε αυτή τη διπροσωπία που μερικές φορές ακολουθούμε σε ό,τι αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για να διδάσκουμε και να κηρύσουμε στα άλλα κράτη-μέλη θα πρέπει καταρχήν να δίνουμε το παράδειγμα. Γι' αυτό λόγο η παράγραφος που αφορά τις, ε, την επιχειρηματικότητα και τις επιχειρήσεις ε, είναι σε συνδυασμό με τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο. Ε, υπάρχουν πολλές ανησυχίες σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό του εμπορίου σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η δύναμη των δυνάμεων. θέλουμε να είμαστε μια ανθρώπινη δύναμη όμως γιατί αυτό προσδοκούν τόσοι πολλοί από εμά. Και να συγχαρώ και τον κύριο Λαμπρινίδη για την εξαιρετική, εξαιρετική δουλειά που κάνει και για την ανανέωση τη θητεία του. Ευχαριστώ. <coughs> Euh, vreau să vă anunț imediat. Vreau să vă anunț că într-o θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ και εγώ και θέλω να επισημάνω ότι ήδη έχουμε χρονική καθυστέρηση. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους ε, συναδέλφους να μην υποβάλουν μπλε κάρτες γιατί έτσι κι έχουμε καθυστερήσει. Τώρα λοιπόν το λόγο έχει ο κύριος ε, Ντέμερ για 1,5 λεπτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η έκθεση, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ένα έργο το οποίο περιγράφει πάρα πολλέ εξελίξει ε, και συγχαίρουμε το συντάκτη. Ορισμένε εξελίξει είναι θετικέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον αρκετά εργαλεία για να εφαρμόζει πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όμω μερικέ φορέ θα πρέπει ε, σε αυτά τα εργαλεία να προσθέσουμε και την βούληση. Σε κάποιε περιοχέ, στην Νότια Αμερική παραδείγματο χάνει, υπάρχει πρόοδο, αλλά σε άλλε η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ακόμα χειρότερη. Η Ρωσία, που αναφέρθηκε σήμερα επανειλημμένα, είναι δυστυχώ μία από αυτέ τι δυσάρεστε περιοχέ. Η Ρωσία πλέον αποτελεί για μας στρατηγική πρόκληση και θέλω να σας παραπέμψω στο ψήφισμα σχετικά με την ανησυχητική κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κρυμαία. Οι Τάταροι είναι ένας ε, μικρός λαός, πολύ περήφανος όμως. Ε, το παρελθόν τους ε, είναι κάπου σκοτεινό, είχαν εκτοπισμούς, διακριτική μεταχείριση βάρους τους, αλλά η Κρυμαία είναι η πατρίδα τους και ήταν παντερίνικη. Σήμερα δεν μπορεί να κάνει κανείς λόγο για ανεκτικότητα στην περιοχή αυτή. Πολλές οργανώσεις έχουν επισημάνει ότι υπάρχουν διακρίσεις εις βάρος των Τατάρων της Κρυμαίας, οι οποίοι δεν έχουν καμία υγειονομική περίθαλψη και δεν θα την ε, έχουν ε, αν δεν κρατήσουν το ουκρανικό σε διαβατήριο. Πρέπει να προστατεύσουμε και άλλους, παραδείγματο χάρη τις θρησκευτικέ μειονότητε στη Μέση Ανατολή. Πάντως την Κρυμαία ένα χρόνο μετά την προσάρτησή της δεν δικαιούμεθα να την ξεχνάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενη μιλήτρια για δύο λεπτά. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Παντσέρη για την έκθεσή του που είναι υπόδειγμα έκθεσης που δεν αποκλεί, γιατί έχει περιλάβει όχι μόνο τις, κοινο... τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αλλά περιλάβει και πολλές ανησυχίες που ταλανίζουν όλους μας. Επίσης είναι αξιοσημείωτη η διαπίστωση ότι η ατιμορρησία θα πρέπει να παταχθεί, να στηρίξουμε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των γυναικών, των παιδιών, των ΛΟΑΔΜ και επίσης να αναφερθώ και σε κάτι άλλο, την ανάγκη να προασπίσουμε τους υπερμάχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί έρχονται στο Κοινοβούλιο, μας διαφωτίζουν, μας εμπνέουν και μετά επιστρέφουν στις θέσεις τους ε, όπου είναι εκτεθειμένοι σε κίνδυνο. Μια, ε, σε ένα από τα 215 εκτιμώντας τις αιτιολογικές σκέψεις ε, αφορά την πρόσβαση σε πόσιμο είδωρ και την πρόσβαση σε, στην αποχέτευση. Αυτά είναι θεμελιώδη δικαιώματα που το 2010 έχουν αναγνωριστεί στα Ηνωμένα Έθνη. Τα δεχόμαστε όλα αυτά, αλλά δεν τα τηρούμε. Είναι αδιανόητο. 15% του παγκόσμιου πληθυσμού, δηλαδή 1 δισεκατομμύρια άνθρωπα, δεν έχουν πρόσβαση σε μία τουαλέτα. Πρέπει να κάνουν τις ανάγκες τους στην ύπεθρο. Ενώ κάθε δύο λεπτά ένα παιδί χάνει τη ζωή του από διάρρεια. Μπορούμε να προλάβουμε την ε, διάρρεια, τον τύφο, την υπατήτηδα. Ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πρόσβαση στην αποχέτευση, γιατί ε, η, ανάγκη να κάνει κανείς την ανάγκη του στην ύπεθρο είναι βάρος της ανθρώπινης υγείας και θα ήθελα να στηρίξω την εκστρατεία του Γιάννη Νίλσον που δίνει μάχη ώστε στα Ηνωμένα Έθνη να γενικεύσουμε επιτέλους τον αγώνα αυτό και να έχουμε όλοι δικαίωμα σε αποχέτευση. Η κυρία Βερζιά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως κάθε χρόνο εξετάζουμε αυτή την έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο. Ο κύριος Παντζέριο, εισηγητής μας, αποφάσισε να κάνει ένα, μια έκθεση που να μην έχει διπλά μέτρα και σταθμά. Βέβαια δεν είμαστε άμεμπτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό και δεν μπορούμε να δίνουμε μαθήματα σε άλλους και να κάνουμε κηρύγματα. Επίσης, μεγάλη θέση δίνεται στην, Ευρωπαϊ... στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και στα κοινωνικά δικαιώματα. Γιατί όμως να μην ε, θεσπίσουμε ένα παγκόσμιο δεσμευτικό μηχανισμό για να σταματήσουμε την ατιμορρησία των μεγάλων πολυεθνικών, γιατί να μην καταδικάσουμε την... Ε, τον ολέθριο αντίκτυπο των ε, σχεδίων προσαρμογής ε, στα κοινωνικά δικαιώματα. Δεν μπορούμε να μιλούμε απλώς ε, ανεπιφύλακτα για τη συνεργασία με τρίτες χώρες σε θέματα μετανάστευσης και να ξεχνούμε ε, τι γίνεται στη διαδικασία του Χαρτούμ και τη συνεργασία με τους δικτάτορες του κέρατος Αφρικής. Επίσης, το παράρτημα για, τα ανθρώπινα, για τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων μου δημιουργεί πρόβλημα γιατί είναι πολύ περιοριστικό και επίσης έτσι σε κίνδυνο όσους παραλείπονται από το παράρτημα αυτό. Γι' αυτό και η ομάδα μου, η Γκούε, θα κρατήσει στάση αποχής για την έκθεση. Κυρία Λόχμπιλερ. Πρόεδρε, κυρία Μοργκερίνη, κύριε αξιότιμε κύριε Λαμπρινίδη, η έκθεση που έχει υποβληθεί είναι μια πάρα πολύ καλή παρουσίαση των διαφόρων δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η έκθεση περιλαμβάνει και πάρα πολλές προτάσεις βελτίωσης. Όμω, η έκθεση δείχνει επίση που πρέπει ακόμα να καταβληθούν προσπάθειες, να γίνουν συζητήσεις με διπλωμάτες και οποτεδήποτε γίνονται αυτές ακούμε ότι αυτοί θαυμάζουν ε, τη δική μας ε, την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εν τω μεταξύ όμως ε, ακούμε και κάποιες κριτικέ για τις αντιφάσεις που περιέχει η ευρωπαϊκή πολιτική. Δημιουργούμε στεγανά κάθε χρόνο προκύπτουν πολλοί θάνατοι προσφύγων και όλα αυτά είναι πονίδιστα. Είναι ντροπή το ότι δεν έχουμε βρει ακόμα μια λύση για να υπάρχουν νόμιμες οδοί προς την Ευρώπη και δεν υπάρχει καμία ε, δέσμευση των κρατομελών να δέχονται τους ε, πρόσφυγες. Η έκθεση λοιπόν δείχνει ότι πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν να επιτύχουμε πλειοψηφία και δεν κατέστη δυνατόν να υπάρξει έλεγχος ως προς την ε, συμβατότητα των μέτρων με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως πρέπει να ελέγξει τι μπορεί να κάνει οποτεδήποτε προκύπτουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τι είδους δυνατότητες υπάρχουν για τους ενδιαφερόμενους, για τα θύματα να απευθυνθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει να το θέσουμε στον εαυτό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Κοράου, επόμενος ομιλητής, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας πω ότι και εγώ ε, με ευχαρίστηση διάβασα την έκθεση του κυρίου Παντσέρη. Ήταν μια δύσκολη έκθεση ε, και αρκετά μακροσκελής ε, και εξετάζει διάφορα ειδικά θέματα. Πάντως ε, μου αρέσει πάρα πολύ η προσέγγιση όσον αφορά τον κατάλογο των χωρών ε, που μπορούν να προκαλέσουν ε, πάρα πολλές συζητήσεις. Με πάση περιπτώσει, <clears throat> είναι αλήθεια ότι το σημείο εκκίνησης είναι ε, ασαφές κατά την άποψή μου. Σε μία περίοδο όπου οι εξωτερικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει να ενταθούν με τις τρίτες χώρες για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, προσπαθεί κανείς να παρακάμψει αυτά τα δικαιώματα. Θα έπρεπε να υπάρχουν δεσμευτικές ρήτρε, να υπάρχουν αποτελεσματικοί έλεγχοι. Γιατί εντάξει υπάρχουν τα ψηφίσματά μας, αλλά ίσως και να μην γίνονται και απόλυτα σεβαστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενος, ε, κύριος, ε, η κυρία, η κυρία Ντότζ Νταϊάνε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η έκθεση ε, αναδεικνύει πολλές ε, τη ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντίον παιδιών, γυναικών, κοριτσιών, ε, κατά της, ε, του θρησκεύματο, του δικαιώματο, της συνεταιριστέ κλπ. Ορισμένες φορέ νιώθουμε ότι όλα αυτά είναι πολύ μακριά, αλλά στη Βόρεια Ιρλανδία στι 26-27 του μηνό, το Δημοσίου Σωματοδοτούμενη Επιτροπή Ισότητας θα ε, αντιμετωπίσει το δικαστήριο την Ushers, μια ε, ε, εταιρεία, μικρή εταιρεία η οποία αρνήθηκε να φτιάξει ένα γλυκό με ένα μήνυμα υπέρ του γάμου των ομοφιλοφίλων. Ε, τέτοιου είδους πράξεις είναι πραγματικά ε, καταπάτηση του άρθρου 9 των, της Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ε, οι νομοθέτες λοιπόν είναι όπως είπε η δικαστής μας η Lady Hill, μια ε, εύλογη ε, ε, ρύθμιση για τους ανθρώπους που, ε, που έχουν αυστηρές θρησκευτικέ πεπιθήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να στείλουμε αυτό το μήνυμα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζιμπ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση με θέματα ανθρώπινα δικαιώματα ε, και κυρίως αιτήσια έκθεση είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα και είναι πολύ δύσκολο να μείνουν όλοι ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή, τον κύριο Πατζέρη, για την εκπόνηση της έκθεσης. Ε, το έτος 2013 είναι ε, χρόνος έναρξης δύσκολων αλλαγών για την Ουκρανία. Έχαμε τα γεγονότα στο Μαϊντάν, πολλά θύματα. Επίσης, πολλές αλλαγές μετά την την Αραβική Άνοιξη. Υπάρχει πρόβλημα με την ε, γαλλική διερμηνία. Please continue. Okay. Thank you. Ε, Συνεχίστε κύριε Ξύπ. Το 2013 είναι και η έναρξη τραγικών δραματικών αλλαγών στην Εγγύη Ανατολή. Ε, και έχουμε πολλά θύματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, εξαιτία ε, της προέλασης του αυτοκαλούμενου Ισλαμικού κράτους. Έχουμε ε, ε, τις ιστορικές επιθέσεις σε πολιτιστικά χριστιανικά αγαθά στην πόλη Μαλούλα στη Συρία, δολοφονίες μειονοτήτων, αναγκαστικούς προσιλητισμούς. Είχαμε πολλές τέτοιες εγκληματικές ενέργειες Επίσης, ε, επιδεινώνεται η κατάσταση των χριστιανών ε, σε όλο τον κόσμο, αλλά και των ε, πιστών άλλων κοινοτήτων. Στην Βόρεια Κορέα, στην Αφρική, είχαμε πάνω από 100 εκατομμύρια χριστιανούς που διώκονται στον κόσμο και χιλιάδες είναι οι χριστιανοί που χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο. Έχουμε τέτοια γεγονότα που φυσικά πραγματώνονται στα πλαίσια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αφρική, στο Μάλι, στο Σουδάν, στην Ιγυρία, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Αυτές είναι οι αρνητικές εξελίξεις, αλλά είχαμε και θετικές εξελίξεις, όπως είναι η έναρξη το 2013 της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία ή η απονομή του βραβείου Ζαχάροφ, που διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο επιβραβεύοντας ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δύο λεπτά. Ο κύριος Βάιντεν Χόλτσερ. Ο κύριος Παντσέλη παρουσίασε μια φιλόδοξη, φιλόδοξη έκθεση, εστιάζει την προσοχή του στα βασικά θέματα και με τον τρόπο αυτό αποφεύγει το λάθος ε, του να απαριθμεί λάθη και με τον τρόπο αυτό η έκθεση δεν μπορεί να δεχθεί, επειδή είναι ακριβώς γενική, πάρα πολλές επιθέσεις. Το Κοινοβούλιο λοιπόν ε, έχει τη δυνατότητα να αντιδρά με ταχύτητα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ συστήνω αυτό που λέει η έκθεση, το να συσταθεί μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία συστηματικά θα επιλαμβάνεται μιας ε, ακριβούς ε, έρευνας κυρίως στο χώρο των ακτιβιστών πρέπει να υπάρχουν κάποια στάνταρτ στην πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν δεν υπάρχουν, αυτό αντιβαίνει με την ε, πολιτική, εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να υπάρχει οπορτουνισμός. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί, δεν υπάρχουν ε, σημαντικοί και λιγότερο σημαντικοί ε, εκπρόσωποι και περιπτώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το να εκφράζει κανείς ε, προειδοποιήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτό είναι επένδυση στο μέλλον. Μόνο αν υπάρχει κράτος δικαίου, αν ισχύουν η δημοκρατία και η ελευθερία, μόνο τότε ζούμε σε έναν ασφαλή κόσμο. Μια τέτοια λοιπόν πολιτική δεν μπορεί να είναι από αλλά θα πρέπει μια τέτοια πολιτική να είναι το αποτέλεσμα συνεργασίας. Ο θεσμός του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, του κ. Λαμπρινίδη, που επιτελεί το έργο του με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα, αυτός ο θεσμός είναι πολύ σωστός και πρέπει να επεκταθεί και να ενισχυθεί περαιτέρω. Επόμενος ομιλητής παρακαλώ. Ο κύριος Μπέλτερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η έκθεση Παντσέρη είναι πολύ ρητή στην ε, καταδίκη των όσων καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και θα πρέπει να εφαρμόσουμε το ψήφισμα περί θρησκείας. Παράγραφος 132 μιλάει για ευρωπαϊκές κατευθύνσεις γραμμές και την προστασία του, της ελευθερίας του θρησκεύματος. Δεν έχουν γίνει και πολλά πράγματα όμως σε ό,τι αφορά την εφαρμογή αυτών των κατευθύνων γραμμών. Θα ήθελα να ρωτήσω τι έχει γίνει ακριβώς. Υπάρχει μια έλλειψη πολιτική βούληση. Εμεί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχουμε έλλειψη πολιτική βούληση, αλλά χρειαζόμαστε πολιτική βούληση και αλλού. Συμφωνείτε λοιπόν με αυτή την αρχή. Ευχαριστώ. Mr. Chairman, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι υποτίθεται προϋπόθεση για τις ε, σχέσεις μας με τρίτες χώρες. Όμως, ε, οι χώρες, για τις χώρες οι οποίες παραβιάζουν το, το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα ή ε, που έχουν ε, καταλάβει ξένες περιοχές υπάρχει κάποιο, κάποια ποινή. ο Πρωθυπουργό του Ισραήλ της προάλλης είπε ότι δεν υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών. Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. η Αρμενία, ε, ε, εκπρόσωπος της Αρμενίας είπε τις προάλλες ότι η, Ρωσία είναι βασικός ε, σύμμαχος στην οικονομία και στο στρατικό τομέα και ότι η Ρωσία αποτελεί εγγύηση για την ασφάλεια της χώρας του. Επίσης η κυβέρνηση του Μαρόκου, ε, εταίρος μας εξίσου, πολύ σύντομα διοργανώνει στην Τάλα ένα συνέδριο. Ντάλα ε, είναι ένα μέρος το οποίο έχει καταλάβει το Μαρόκο εις βάρος της Δυτικής Σαχάρας. Ε, θα αλλάξουμε κάτι κυρία Μογκερίνη σε ό,τι αφορά την ε, πολιτική μα σχέση με αυτές τις χώρε. Ο κύριος Τερικάβρας, ένα λεπτό. Είναι αλήθεια ότι την τελευταία δεκαετία η θέση των γυναικών στην κοινωνία έχει υποστεί εντυπωσιακή βελτίωση. Παρ' όλα αυτά, κοινωνικές, ε, πολιτικές και πολιτιστικές ανισότητες μεταξύ άνδρων και γυναικών εξακολουθούν να επιβιώνουν ακόμη και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να σας παραθέσω ε, κάποια γραπτά του John Stuart Mill πριν από 146 χρόνια. Και μάλιστα εκεί μιλώντας για τις γυναίκες λέει ότι το όφελος ε, που θα αποκτήσουμε ε, χειραφετώντας τις γυναίκες και αφήνοντας, την αφήνοντας ελεύθερη επιλογή του επαγγέλματός τους και προβλέποντας ε, ίδια αμοιβή για ίδια εργασία όπως τα υπόλοιπα ανθρώπινα όντα, το όφελος θα ήταν να διπλωσιάσουμε το δυναμικό των διανοητικών ικανοτήτων προς όφελος της ανθρωπότητας. Πριν από 146 χρόνια διατυπώθηκε μια τέτοια έκκληση και ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο... Ένα λεπτό. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Πατιστέλη καταδικάζει τους ε, ε, συνδικαλιστές ε, για την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης υπάρχουν κατηγορίες σχετικά με διακριτική μεταχείριση κατά ε, εκείνων που δεν ε, προσλαμβάνουν περισσότερο προσωπικό. Αυτά όλα είναι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εργαζομένων, όμως η Ολλανδική κυβέρνηση δεν επιτρέπει την εφαρμογή της απόφασης. Και αυτό που πραγματικά μας σοκάρει είναι ότι η ΥΠΟΛ όχι μόνο μοιάζει είναι πάνω από τον θεσμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και πάνω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να ζητάμε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν εμείς επιτρέπουμε να υπάρχουν τέτοιε παραβιάσεις μέσα σε ένα οργανισμό και αυτό μάλιστα εξ ονόματο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Σοπραντ για ένα λεπτό. Η έκθεση Παντζέρη καταδεικνύει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν, ε, αποτελούν πλέον εξωτερική πολιτική. Ε, έχουν ζητούμε από τα κράτη να καταλήψουν την εθνική τους εξωτερική πολιτική ε, και να ακολουθούν απλώς μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει απλώς ισχύ στο, στη διεθνή σκηνή, δεν θέλει να είναι ένας από τους πολλούς πόλους, ε, θέλει απλώς να εξάγει ε, την ε, κουλτούρα του, τρόμου τρόμ και του, φόνου με την πρόθεση των αμβλώσεων και την, τον πόλεμο κατά της φυσικής οικογένειας. η το δηλητήριο της ακροδεξιάς ε, ε, διαλύεται σε μικρότερες δόσεις ε, μέσω της, των κατηγόρων που ευθύνονται εναντίον της Κίνας και της Ρωσίας. Όμως αυτοί που ξέρουν και είναι υπερασπιστές του δικαιώματος της ζωή θα ψηφίσουν εναντίον της έκθεσης Παντσέρη. Ο Κύριε Πρόεδρε, το Συμβούλιο ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Πλαίσιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία προκειμένου να ενισχύσει τις σχέσεις μας και τη δέσμευσή μας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και έχουμε και ειδικό εντεταλμένο για τα ανθρώπινα δικαιώματα για να καταστήσουμε πιο αποτελεσματικό το έργο μας. Τώρα έχουμε καλύτερα μέσα για να ε, προασπίσουμε από κοινού τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο. Παρ' όλα αυτά δίνουμε μάχη και μερικές φορές ε, πασχίζουμε για να διατρανώσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί μερικές φορές διαφωνούμε και μεταξύ μας και είναι κρίμα που μια τέτοια έκθεση χρησιμοποιείται ε, ανάρμοστα και εγωιστικά από ορισμένους ευρωβουλευτές για να ενισχύσουν την εσωτερική διχόνοια για θέματα που αποτελούν αποκλειστικές εθνικές αρμοδιότητες. Είναι ακατάλληλη αυτή η συμπεριφορά και θίγει την αξιοπιστία μας. Θα πρέπει να πατάξουμε κάθε τέτοια προσπάθεια που ε, ξεφεύγει από θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ε, παραβίαση των ε, δικαιωμάτων γυναικών και παιδιών, μειονοτήτων, της διώξης των χριστιανών και ούτω καθεξής. Ο κύριος Χάουιτ, για 1,5 λεπτό. Συγγνώμη, η ε, κυρία Βαλενσιάνο, όχι μπλε κάρτα ελπίζω. Όχι μπλε κάρτα, διαδικαστικό κύριε Πρόεδρε. Γιατί μπορεί να οφείλεται στη διερμηνία το πρόβλημα, γιατί ο προλαλής σας, ο προηγούμενος ομιλητής, μίλησε για τους ΛΟΑΔ, ομοφιλόφιλους, λεσβίες, ε, ε, διαφιλικούς και φιλομεταβατικούς, τους χαρακτήρισε δηλητήριο αν δεν ήταν λάθος η διερμηνία, θα παρακαλούσα τον συνάδελφο να ανακαλέσει. Δεν μπορεί κανείς να χαρακτηρίζει τους ομοφιλόφιλους δηλητήριο της κοινωνίας. Είναι απαράδεκτο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, ε, e, Σαν μπλε κάρτα μου ακούγεται αυτό που είπατε, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δώσω το λόγο στον Ρίτσαρντ Χάουιτ για 1,5 λεπτό. Θα χρησιμοποιήσω το χρόνο μου για να εστιάσω σε ορισμένες ε, πτυχές της έκθεσης σε ό,τι αφορά τις κατευθύνσεις γραμμές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Λαμπρινίδη για την προσωπική του στήριξη σε αυτό το θέμα. Η Ευρώπη δημιούργησε ε, την ιδέα των εθνικών προγραμμάτων δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα που υιοθετήθηκε από τον πρόεδρο Ομπάμα. Ελπίζω όλα τα κράτη-μελή θα ε, το υιοθετήσουν και θα ολοκληρώσουν τα σχέδιά τους. Και, και ότι θα δείτε τη συνολική εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων εσείς. Θα χρειαζόμαστε όμως και ευρωπαϊκές συστάσεις για το πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να ασκούν τη δέουσα επιμέλεια σε ό,τι αφορά την, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, πλέον έχουμε συγκεκριμένες ε, υποχρεώσεις ε, υποβολής εκθέσεων ε, και θα ήθελα η ύπατη εκπρόσωπος να αναλάβει την εφαρμή αυτού του πλαισίου και να στηρίξει και τον κύριο Μπάνκι Μουν στις προσπάθειές του όλο αυτό, όλες αυτές οι υποχρεώσεις να γίνουν παγκόσμιες και όχι να περιοριστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να διευκολύνουμε την πρόταση στη δικαιοσύνη ανθρώπων που είναι θύματα ε, της ε, ε δράσης που αντιβαίνει στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο κύριος Γιούρεκ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή που έπρεπε να μιλάει για, ε, για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μερικές φορές ε, ε, ξεφεύγει από αυτό το θέμα. Στο σημείο 65 ε, γίνεται μια ολόκληρη επίθεση στην, στην βούληση ολόκληρης κοινωνίας των Κροατών και των Σλοβακών. Μιλάει η παράγραφος 165 κατά του δημοψηφίσματος στις δύο αυτές χώρες που τάχθηκε στον περιορισμό του γάμου μόνο σε, στα δύο φύλλα. αν εμείς σήμερα ε, ασκούμε επίθεση ολόκληρους λαούς που έχουν αποφανθεί μέσω ενός ε, δημοψηφίσματος και τάσσονται υπέρ μια συγκεκριμένη μορφή οικογένειας, τότε πώς ε, θα προστατεύσουμε ανθρώπους που υφίστανται μονομένα επιθέσεις γιατί το κάνει υποτίθεται στο, στο όνομα της ομοφοβίας και όμως και η, η Πολωνική Βουλή ε, είπε με σαφήνεια ότι ακριβώς επειδή ε, πρεσβεύει τις ε, ιουδεοχριστιανικές αξίες δεν μπορεί να δεχτεί κάποιες, κάποια ευρωπαϊκά κείμενα που αναφέρονται στην ομοφιλοφοβία. Η κυρία Φεράρα. Ως ε, εισηγήτρια για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλω να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα την έκθεση του συναδέλφου κυρίου Παντσέρη. Ε, πρόκειται για την αμφισβήτηση των θεσμών και του θεσμικού πλαισίου στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι στα θεμελιώδη δικαιώματα ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε αναλάβει να είναι ο εγγυητής του χάρτη των θεμελιωτών δικαιωμάτων. Η ύπατη εκπρόσωπος, η κυρία Μογκερίνη, επίσης έχει αναλάβει αυτό το ρόλο. Άρα δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει ε, σεβασμός από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να επιμείνουμε στην επιδίωξη εφαρμογής και επίτευξης αυτών των στόχων. Γι' αυτό λοιπόν εγώ προσωπικά θα ήθελα να προτείνω ότι πρέπει να υπάρχει μια εσωτερική στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα που είναι συνεπής με το στρατηγικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και όλα αυτά και στις εξωτερικές μας σχέσεις. Επίσης να μην υπάρχει το δίλημα της Κοπενχάγης. Να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά το κράτος δικαίου και αυτό όχι μόνο ε, για τα κράτη πριν από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τα ίδια τα κράτη-μέλη. Ο κύριος Βόικτ επόμενος ομιλητής για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, γίνεται πολλή λόγος ε, για την καθοριστική σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο οι τρίτες χώρες. Θα πρέπει να ασχολούμεθα και με την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα ίδια τα κράτη-μέλη. Κατά νου έχω την Πολωνία και τη Ρουμανία. Ε, μήπως ε, εκεί δεν θέλουμε να ξέρουμε ότι βασανίζονται άνθρωποι. Μήπως υπάρχουν και άλλες χώρες που να υπάρχουν παρεμβάσεις ε, στην Αυστρία μετά από 60 χρόνια σε μία σύμβαση αναφέρεται ότι οι άνθρωποι μπορούν να φυλακιστούν μέχρι και 15 χρόνια όταν εκφράζουν την άποψή τους. Στη Γερμανία άλλοι 13 βρίσκονται σε δικαστικές διαμάχες λόγω ελεύθερης άποψης, έκφρασης άποψης. Εξάλλου ε, υπάρχει και περίπτωση όπου κάποιος βρίσκεται στη φυλακή για 12,5 χρόνια και πολύ γρήγορα θα πρέπει να πάει στο ψυχιατρίο. Επτά ευρωβουλευτές εδώ και 18 μήνες είναι στη φυλακή χωρίς καν να τους έχει απευθυνθεί κατηγορία. Στην Ελλάδα αυτό. Πώς γίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. διαπιστώνω ότι έχουν γίνει δεκτές οι προτάσεις μου για τα δικαιώματα των εθνοτικών, θρησκευτικών και άλλων μειονοτήτων στην έκθεση. Γιατί οι ειδικέ περιστάσεις ε, χρήζουν ειδικών λύσεων για να εξασφαλιστεί ισότητα δικαιωμάτων. Βέβαια, οι πιο δύσκολε καταστάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντοπίζονται στη Μέση Ανατολή με τι διώξει των χριστιανών και κυρίω γυναικών και παιδιών που ε, συνελήφθησαν, απήχθησαν, βασανίστηκαν ή κατέστησαν σκλάβοι εξαιτίας των θρησκευτικών πεπιθήσεών τους. Είναι απαράδεκτες διώξεις πιστών θρησκειών. Δεν μπορούμε να μένουμε σταυρωμένα χέρια μπροστά σε τέτοια φαινόμενα κατάφορης παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι πραγματικά εγκλήματα αυτά που διαπράττονται εις βάρος των χριστιανών. Θα πρέπει να βρεθούν κάποιοι μηχανισμοί να μπορέσουμε να αντιδράσουμε σε αυτά τα εγκλήματα. Σας είχα ανακοινώσει από την αρχή ότι δεν επιτρέπονται παρεμβάσεις με μπλε κάρτα, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Κύριος Κρίστε, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω τη συγχαρητήριά μου στον άλφο κύριο Παντσέρη για αυτή την ιδιαίτερα ισόρροπη έκθεση και για τον επαγγελματικό τρόπο με τον οποίο τη συνέταξε. Με την ευκαιρία της διεθνού ημέρα ε, γυναικών θα ήθελα και εγώ να εκφραστώ για τη βία που ασκείται εις βάρος των γυναικών ε, για περιπτώσεις εξαναγκασμού σε άμπλωση και θα ήθελα να μιλήσω και για την παιδική εργασία. Αυτές είναι, είναι οι δεχτή εγκλήματα. Το Γαλλικό Ινστιτούτο για τη Δημοκρατία δημοσίευσε μια σχετική έκθεση και αναφέρει ότι η επιλεκτική άμβλωση αυτή μπορεί να επεκταθεί και να αφορά και χώρες στα Βαλκάνια και στην Κεντρική Ασία όπου υπάρχει ανισορροπία ανάμεσα ε, στα γόρια και τα κορίτσια. Και αυτό που έχει επίσης σημασία είναι στις κατευθυντήριε γραμμές τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη βία ει βάρο των γυναικών και των κοριτσιών να συμπεριλάβουμε και το θέμα της επιλεκτικής άμβλωσης. Χρειαζόμαστε δείκτες, χρειαζόμαστε δεδομένα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Όσον αφορά τώρα την παιδική εργασία, πράγματι υπήρξε πρόοδος και θέλω να σας επισημάνω ότι είναι δική μας δουλειά, δουλειά των Ευρωβουλευτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο πλαίσιο που να μην υπάρχει παιδική εργασία. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τόμασιτς έχει το λόγο. Για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Είμαι γενικώ υπέρ τη έκθεση, αλλά ω ε, Ευρωβουλευτή από την Κροατία θα ήθελα, αισθάνομαι το καθήκον να αντιδράσω στην παράγραφο 165 τη ηθίκη, όπου ο εισηγητή εκφράζει τη λύπη του για την έκβαση του κρατικού δημοψηφίσματο για τον ορισμό του γάμου από το Δεκέμβριο του 2013. Θεωρώ ότι δεν έχει λόγο να λυπάται ο εισηγητή, γιατί ο συνταγματικό ορισμό του γάμου στην Κροατία που δεν φύγει τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ. Αντίθετα, αποτέλεσε κατα... καταλήτη για την έγκριση του νόμου για, το σύμφωνο συμβίωση μεταξύ ανθρώπων του ίδιου φύλου του Ιουλίου του 2014. Ε, γιατί πιστεύω ότι κάθε κοινωνία πρέπει να μεριμνά για όλα τα μέλη της και η επιθυμία ε, των Κροατών, της ε, πλειοψηφίας τους, να είναι ο γάμος ένωση ενός άνδρα και μιας γυναίκας, δεν είναι έκφραση ομοφοβίας ή διάκρισης όπως υπενήσεται η παράγραφος 125. Αντίθετα, αποτελεί έκκληση για την προστασία παραδοσιακών αξιών που κράτησαν ομοιογενή την κοινωνία μας ε, όταν συνταραζόταν από συχνές ιστορικές αντιξότητες. Σας ευχαριστώ. Ο Χτες ε, ψηφίσαμε την έκθεση Ταραμπέλα, Βέλγου σοσιαλιστή, που η κυρία Grip ε, συνεχάρει εκ μέρους του ΕΛΚ. σήμερα είναι η ώρα ενός άλλου σοσιαλιστή, του κυρίου Παντζέρη, την οποία θα υπερψηφίσουν πολλοί από το ΕΛΚ. Εγώ ψήφισα εναντίον του Ταραβέλα και θα ψηφίσω και εναντίον της έκθεσης Παντζέρη, εξαιτία του ότι προωθεί μια επικίνδυνη ιδεολογία η ιδεολογία η οποία προωθεί, ε, κοινοτικοποιεί κάποιες ε, μειοψηφικές απόψεις. Θέλουμε να επιβάλλουμε τα, τη δική μας θεώρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο, ενώ εμείς ε, δεν σεβόμαστε ε, ούτε την επιθυμία των λαών, ε, ούτε τις εξουσίες των κρατών μελών. Το ίδιο έγινε και στην Κροατία, που αποφάσισε ο γάμος να είναι μόνο μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτή είναι η δημοκρατία όμως. Ο πρόεδρος διακόπτη. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, έχουμε την 56η επέτειο της εξέγερσης στο Θιβέτ. Εχθές ε, είχαμε σημαίες του Θιβέτ σε 10.000 κτίρια σε πολλές περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά μας υπενθύμησαν την ελευθερία άποψη στα θεμελιώδη δικαιώματα και ότι πρέπει να πάψει να υπάρχει καταπίεση αυτής, ε, της, του, αυτού του ειρηνικού πολιτισμού. έχουμε όλους αυτούς τους Θιβετιανούς που θυσιάστηκαν και πάρα πολλούς ε, που εξακολουθούν να βρίσκονται στη φυλακή. Η τύμπη ομάδα είναι υπέρ του διαλόγου ανάμεσα στους εκπροσώπους του Νταλάη Λάμα και της κινέζικης κυβέρνησης. Το υποτιθέμενο έγκλημα των Θιβετιανών είναι ότι τάσσονται υπέρ των νόμιμων δικαιωμάτων τους, τη διατήρηση του πολιτισμού τους, τη γλώσσα τους, τον πολιτισμό τους. Εμείς λοιπόν θέλουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε έτσι ώστε επιτέλους να πάψει να υπάρχει αυτή η ταπείνωση του θηβετιανού λαού. Η κυρία Ροντρίγκης για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ την ε, Επίτροπο για το έργο που επιτέλεσε μέχρι τώρα και να πω ότι όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί παντού το σεβασμό της δημοκρατίας, την οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης διέπεται από τις αξίες αυτές, ή τουλάχιστον αυτό θα έπρεπε να γίνεται. Πολλές φορές όμως εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δίνει προνόμια σε αυταρχικά καθεστώτα που παραβιάζουν κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, πολύ εύκολα μπορεί να παραγωνιστεί ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Ιδιαίτερα όταν οι άνθρωποι χρησιμοποιούνται ω ε, όπλα πολέμου. Και πολλέ γυναίκε πέρασαν από την κόλαση αυτή. Γιατί οι γυναίκε εξακολουθούν να είναι το η ασθενέστερη πτυχή του αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να προστατεύουμε τι γυναίκε. Έχουμε το καθήκον να το κάνουμε. Θα πρέπει να ασκήσουμε πολύ μεγαλύτερη πίεση στι εξωτερικέ μα σχέσει με χώρε που επανειλημμένα παραβιάζουν τα στοιχειώδη δικαιώματα και των γυναικών και των ανθρώπων γενικώ. Θα πρέπει επίσης όσοι προσπαθούν να μπουν στην Ευρώπη και κυρίως μετανάστευση γυναικών και παιδιών και ανδρών από την ε, όχθη της Μεσογείου θα πρέπει να προστατεύσουμε και να στηρίξουμε καλύτερα αυτούς τους ανθρώπους για να σταματήσουμε να θεωρούμε ως παράπλευρες ζημιές ε, τους ε, θανάτους στη Μεσόγειο τέτοιες, τέτοιου είδους απώλειες ε, καταφέρουν πολύ μεγαλύτερο πλήγμα στις ευρωπαϊκές αξίες. Ο κύριος Συναδεινός, για ένα λεπτό. Πώς θα χαρακτηρίζατε έναν οργανισμό που διακηρύττει με στόχο τα δημοκρατικά καθεστώτα χαρακτηρίζονται από σεβασμό για το κράτος δικαίου, την ελευθερία του λόγου, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ανεξάρτητη δικαιοσύνη και αμερόληπτη διοίκηση, αλλά όταν του καταδεικνύουν ότι ένα από τα μέλη του παραβιάζει κατάφορα τις προαναφερθείς αρχές λόγω πολιτικών σκοπιμοτήτων, εθελοτυφλοί σε αυτόν τον χώρο είχαμε επισημάνει με στοιχεία την παρέμβαση της τότε φασιστικής συγκυβέρνησης αλλά και του ίδιου του πρωθυπουργού σαμαρά στην υποτιθέμενη ελληνική τυφλή δικαιοσύνη για τη σύλληψη του αρχηγού βουλευτών και μελών της χρυσής αυγής της τρίτης εκλογικά δύναμης και μοναδικής ουσιαστικά αντιπολίτευσης στην ελλάδα. είχαμε ενημερώσει για τις παράνομες διαδικασίες προφυλάκηση χωρίς την άρση Ασυλία και σήμερα εδώ διατυμπανίζουμε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων την προώθηση της δικαιοσύνης τη διαφάνεια την ελευθερία του λόγου. Α ελπίσουμε ότι έστω και αργά θα υπάρξει ενεργό ενδιαφέρον και πίεση στην ελληνική κυβέρνηση για αποκατάσταση δικαιοσύνη και κατ' επέκταση δημοκρατίας ώστε να δοθεί άμεση λύση στην πολιτική δίωξη τη Χρυσή Αυγή. Επίση, ήθελα να προτείνω στην κυρία μογκερίνη να πει στου φίλου τους σκοπιανούς εάν θέλουν να λύσουν τα προβλήματά τους θα ενωθούν με την ελλάδα. Ο κύριος Ντάβορ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ σημαντικό μέσο για τον προσανατολισμό τη εξωτερική μα πολιτική και τη πολιτική συνεργασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε στα κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω να διαγραφούν τελικά από το ψήφισμα ε, κάποιε μνήε ε, στα κράτη-μέλη. Δεν έχουν τη θέση του εδώ. Επίση, ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το χάρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών γιατί μερικές φορές γίνεται ο χάρτης αυτός μέσω κάποιων ιδεολογικών αγώνων και αντιπαραθέσεων. Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα και ξέρουμε ότι ε, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ξεκινά και πριν από, την, από τη γέννηση, ήδη από την εμβριακή φάση. Επίσης, οι ε, ίδιες αρχές θα πρέπει που εφαρμόζουμε ε, για τα κράτη-μέλη θα πρέπει να τις σεβόμαστε και με τις τρίτες σχέσεις. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε σε τρίτες χώρες πράγματα που δεν εφαρμόζουμε εμείς. Γιατί μερικές φορές το κύμα, το έβριο το θεωρούμε ως απλό απόρριμα που το πετάμε. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την προστασία της ζωής και όχι μόνο την προστασία του δικαιώματος του θανάτου. Κύριε τα δύο μέτρα και δύο στάθμα ε, ε, αφήνουν ε, ατιμόρυτους ε, πολλούς ε, από αυτούς που παραβαίνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα για να αποτελούν μαχαιριά στην πλάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι σχέσεις με τρίτες χώρες μέσω της αναπτυξιακής βοήθειας θα πρέπει να περνάνε από μια επίσκεψη σε αυτές τις χώρες να δούμε ποιοι είναι στις φυλακές τους. Πολλές χώρες με τις οποίες έχουμε ειδικέ σχέσεις φυλακίζουν ακτιβιστές, bloggers, δημοσιογράφους κλπ ε, και ελέγχουν ε, την δικαιοσύνη έτσι ώστε να καταπιέζουν τους ανθρώπους αυτούς. Ε, εμείς εστιαζόμαστε στους διμερείς διαλόγους, αλλά αυτό δεν είναι λύση, γιατί δεν χαρακτηρίζεται το διμερείς διάλογος από διαφάνεια ε, και γι' αυτό το λόγο αποτυγχάνουν. Το Συμβουλίο Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση το σύνολό της, θα πρέπει να επενδύσει σε ε, πολιτικές που θα έρθουν κοντά στους πολιτικούς ακτιβιστές και θα ε, ελέγχουν την ε, συμπεριφορά των κρατών με τις οποίες, με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Πάρτε την Αιθιοπία και άλλες χώρες θα έπρεπε να ζητάμε, για παράδειγμα, να απελευθερώνουν όλους τους ε, πολιτικούς ε, ε, κρατούμενους που έχουν, προκειμένου να συνεργαστούν μαζί τους. Ο Ευρωπαϊκό Εντάλμενο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει εργαστεί πολύ σωστά. Ο πρόεδρο διακόπτει την ομιλήτρια δυστυχώ. képviselő asszony pontosan Μιλήσατε 30 δευτερόλεπτα παραπάνω από όσο επιτρεπόταν. Ε, παρακαλώ πολύ προσέξτε το. Θα ζητήσω από τους συναδέλφους ε, να σέβονται το χρόνο τον οποίος έχει δοθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ο μεγάλος Ρώσος ε, ανθρωπιστής Σαργκέ Κιόγελοφ ε, κάποτε προτάθηκε για το βραβείο Νομπέλ Ειρήνης κατά τη διάρκεια του τσετσενικού πολέμου όπου οι Ρώσοι δολοφόνησαν ε, χιλιάδες ανθρώπων σε Τσενία, Κοβάλη είπε «Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορεί να είναι εσωτερική υπόθεση μόνο μίας χώρας». Το γεγονός λοιπόν ότι δεν έλαβε το βραβείο Νομπέλ, αυτό κατ' ουσίαν έδειξε και απέδειξε ότι τα τελευταία χρόνια η πολιτική είναι αδιάφορη απέναντι στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θεωρούν ότι ε, απλά είναι θέμα δικαιοσύνης και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σιγά σιγά πολλοί πιστεύουν ότι δεν είναι απαραίτητο να προστατεύονται οι πιο αδύναμοι. Τα εμπορικά συμφέροντα επικρατούν. Η έκθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιβεβαιώνει αυτό που είπε ο υποψήφιος νομπελίστας ότι δηλαδή παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορεί να είναι μόνο εσωτερική υπόθεση μιας και μόνο χώρας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα λοιπόν, ε, επόμενος... Ε, Μιγιάν Μον, ε, ευχαριστώ. Η ετήσια έκθεση που συζητούμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα δείχνει πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι από τα σήματα κατά τεθέν μα. πολύ σημαντικό στοιχείο τη ταυτότητά μα και θα πρέπει να έχει ιδιαίτερη θέση και στην εξωτερική μας πολιτική. Ιδιαίτερα μια στιγμή που αφισβητούνται κάποιες διεθνείς αξίες και μάλιστα αναδεικνύονται κάποια εναλλακτικά μοντέλα πολιτικής οργάνωσης. Έχουμε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο με πολλές κρίσεις και προβλήματα και μάλιστα πολλά τέτοια βλέπουμε και στις γειτονικές μας χώρες ε, και προς Ανατολάς και προς τον Νότο. Έχουμε πολλά παραδείγματα κατάφορων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκεί και με βάση το άρθρο 8 της ε, συνθήκης θα θέλαμε η ζώνη της γειτονίας να έχει ως θεμέλιο ακριβώς ε, τις αξίες μας και μία από αυτές είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η πολιτική γειτονία ε, χρήζει μέσων και μέσω και μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων και φυσικά χρήζει και ρεαλισμού. Δεν μπορούμε να ξεχνούμε στην πολιτική αυτή τις αξίες μας. Επίσης, ε, σημαντική είναι η ανάγκη εξωτερική δράση να λαμβάνει υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί η ειρήνη και η ασφάλεια, ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι τα σύνθημα των αρχών του αιώνα που θα πρέπει να συνεχίσει να μας καθοδηγεί. Ο κύριος Ρανζέλ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, καλώς ήρθατε, κυρία Μοκερίνη. Η πρόταση, θα ήθελα μάλλον να εστιάσω την ομιλία μου σε δύο πράγματα. Πρώτον, το θέμα της ε, δημοκρατικής μετάβασης. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί μπορεί να παίξει ένα ρόλο μοναδικό. Ένα ρόλο κρίσιμο, υποστηρίζοντας τις ε, χώρες οι οποίες ε, επιθυμούν να εκδημοκρατιστούν και να υποστηρίξει και τις δυνάμεις μέσα σε αυτές τις χώρες που θέλουν να προετοιμάσουν αυτή τη μετάβαση. Στη Νότια Ευρώπη, στην Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ελλάδα το έχουμε δει στο παρελθόν, αλλά και στην Ανατολική Ευρώπη το είδαμε στο παρελθόν πώς καταφέραμε να επιτύχουμε ε, ειρηνική μετάβαση στη δημοκρατία ε, με προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιστεύω ότι αυτό θα έπρεπε ε, να είναι ένα από τα πράγματα που θα πρέπει να επιστιάσουμε. Δεύτερον, προστασία των κοινοβουλευτικών δικαιωμάτων ως μια σταδιακή διαδικασία. Καμιά φορά είμαστε υπερβολικά απαιτητικοί από χώρες οι οποίες ήδη βλέπουμε ότι κάνουν προσπάθειες. Θα πρέπει να τις βοηθήσουμε. Ευχαριστώ. Κυρία Κομοντίνη, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η έκθεση ε, θίγει πολλά θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά πρέπει να σας πω ότι οφείλουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας εκεί που είναι απαραίτητο να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θέλω να υπάρχει ένα καλύτερο πλαίσιο για την εφαρμογή αυτών των μέτρων, ένα πλαίσιο ε, το οποίο ε, θα προβλέπει την υποστήριξη ορισμένων κρατών στον δρόμο του εκδημοκρατισμού. Τα μέτρα δεν θα πρέπει να είναι μόνο προτεραιότητε, αλλά θα πρέπει να επιδιώκουν συγκεκριμένου στόχου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να είναι συνεπής, να επιδεικνύει ε, συνέπεια τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική πολιτική. Κάτι ε, πολύ συγκεκριμένο. Ε, θα ήθελα να πω ότι η κατακυδεμόνευση των μέσων ενημέρωσης και η υποδιγέτηση ε, κατ' ουσίαν εξυπηρετεί μόνο εκείνους που θέλουν να εκμεταλλευτούν τις χώρες τους και δεν εκφράζει τα συμφέροντα των πολιτών. Γι' αυτό φτάνουμε σε ανθρωπιστικές κρίσεις και αυτό πάλι δημιουργεί τραγωδίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτή λοιπόν την έκθεση αυτό που ενδιαφέρει είναι να δρομολογηθούν συγκεκριμένα μέτρα σε ορισμένα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ κύριο Μπούντα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η ατομική αξιοπρέπεια είναι στοιχεία βασικά που θα πρέπει να διέπουν όλες τις ευρωπαϊκές πράξεις και πολιτικές και να αποτελέσουν και την ύψιστη προτεραιότητα των πολιτικών μας. Δυστυχώς έχουμε ανησυχητική αύξηση ε, της ε, τρομοκρατίας ε, και φτάσαμε στο 62% την τελευταία χρονιά και μάλιστα οι χώρες που έχουν υποστεί τρομοκρατικές υποθέσεις με μεγάλες δολοφονίες πάνω από 50 ατόμων από 15 έγιναν 24. Έχουμε και την απειλή του αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού κράτους στον Αραβικό κόσμο και η ένοπλη σύρεξη στην Ουκρανία. Αυτά είναι λίγα μόνο, λίγα μόνο παραδείγματα των απειλών στην ασφάλεια. Η ασφάλεια είναι σημαντικό θέμα της εξωτερικής μας δράσης και βασικό στοιχείο της ταυτότητάς μας. Θα πρέπει λοιπόν να επισημαίνεται στις διμερείς μας σχέσεις. Ο κύριος... Κούκαν, για ένα λεπτό. Μικρόφωνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το 2013 ήταν ένας κρίσιμος χρόνος σε ό,τι αφορά την ε, απάντησή μας στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Επαναλαμβάνω, θα πρέπει να παραμείνουμε προσιλωμένοι στι αρχέ μα και τι αξίε μα. Αυτό σημαίνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο των σχέσεών μα με τρίτε χώρε. Θα πρέπει η στάση μα να είναι συνεπής και συνεχής με ιδιαίτερη εστίαση στους κοντινού μα γείτονε. Θα πρέπει να στηρίξουμε τι δημοκρατικέ εξελίξει, το κράτο δικαίου και τις ε, ε, ελεύθερε και ανταγωνιστικέ εκλογέ. Αυτά είναι οι βασικές ε, προϋποθέσεις ε, για λειτουργικές ε, δημοκρατίες που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι δυνατόν να υποχωρήσουμε, να συμβαστούμε σε αυτά. Θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτά τα θέματα στη διαδικασία διεύρυνσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Πλέγκοβιτς έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Αντιπρόεδρε, αγαπητέ συνάδελφε Παντζέρη. συζητούμε την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο για το 2013. Και είναι σημαντικό να φανεί από την συζήτηση ότι η αυριανή εκδοχή, η τελική εκδοχή αυτής της έκθεσης θα περιορίζεται στις χώρες που είναι το αντικείμενό τους, δηλαδή στις χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί μιλάμε για την ε, δημοκρατία στον κόσμο. Οπότε παράγραφοι όπως 162 και 165 που είναι επίμαχες αμφιλεγόμενες, ελπίζω να διαγραφούν, να καταπέσουν, δεν έχουν τη θέση τους στην έκθεση αυτή. Και αυτό το λέω όχι μόνο επειδή κατάγομαι από την Κροατία. Είναι πολύ σημαντικό η συζήτηση αυτή επί της έκθεσης συνδυάζεται και με την προηγούμενη μας συζήτηση που αφορούσε την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικές ε, οι ανθρώπινες, οι αξίες μας και οι αξίες για η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην εξωτερική μας πολιτική. Και αυτό είπε ο κύριος Παντζέρη, ότι στις κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει να δώσουμε στι διακοινοβουλευτικέ επιτροπές για τις ε, εργασίες του. τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο. Σας ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κάποιος ε, μίλησε για δηλητήριο στην κοινωνική ζωή αναφερόμενος στην ομάδα στους ΛΟΑΔ. Ε, νομίζω λοιπόν ότι κάτι θα πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί αυτό. Εγώ στη σημειώση που έχω κάνει θα ήθελα να πω ότι χαιρετίζω κυρίως την ελευθερία της ε, θρησκείας, της έκφρασης, ε, την καταδίκη της βίας εις βάρος των γυναικών. Αποδοθεί ιδιαίτερη σημασία στην εξαναγκαστική παιδική εργασία, στην φτώχεια και στην κακή διατροφή. Ακούμε πολλές φρικτές ιστορίες για βιασμό και αρπαγή κυρίως νέων γυναικών. Οφείλουμε λοιπόν να τις βοηθήσουμε και η καλύτερη πολιτική που μπορούμε να εφαρμόσουμε είναι να τις στηρίξουμε, να τις εκπαιδεύσουμε, γενικά να μεριμνήσουμε για την εκπαίδευση. Η έκθεση λοιπόν επαναλαμβάνει τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατία σε όλες τι δραστηριότητε. Τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να είναι στο επίκεντρο όλων των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. Βλέπουμε ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε δεν είναι μόνο λόγια, πρέπει να υποστηρίξουμε την ελευθερία της ε, θρησκείας, της Έκφραση και της σκέψη. Σα ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ε, τώρα λοιπόν ε, περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye και έχουμε 13 ενδιαφερόμενους ε, που έχουν ζητήσει το λόγο. 13 λοιπόν, Σόγκορτ Τσόμποχα έχει καταρχήν το λόγο εκ μέρους του ΕΛΚ. Σας ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, στην έκθεση πολύ σωστά επισημαίνεται το δικαίωμα του συνέρχεστε. Τα κράτη-μέλη πέρα από αυτό καλούνται να ε, καταδικάσουν οποιοδήποτε περιορισμό και περικοπή αυτού του δικαιώματο. Θέλω λοιπόν να σα ενημερώσω ότι σε ένα κρατο μέλο στη Ρουμανία, απαγορεύτηκε μια ειρηνική διαδήλωση μόνο και μόνο γιατί οι πολιτικοί θεσμοί ε, έχουν πρόβλημα με τους πολιτικού στόχου αυτή της ομάδα και αυτής της διαδήλωση, η οποία θα λάμβανε χώρα σε μια μεικτή εθνοτικά περιοχή όπου πριν από κάποια χρόνια είχαμε και εθνοτικέ συγκρούσει. Η περικοπή του δικαιώματος του συνέρχεστε είναι κάτι συνηθισμένο σε ένα αντιδημοκρατικό καθεστώς. Θα έπρεπε λοιπόν να πει κανείς στους Ρουμάνους ότι οφείλουν να αντιμετωπίσουν σοβαρά το πρόβλημα των μειονοτήτων. Γιατί η κατάσταση είναι η εξή. Αρνούνται σε μικρές ομάδες το δικαίωμα, το δημοκρατικό δικαίωμα ειρηνικών διαδηλώσεων. Και νομίζω όταν κάτι τέτοιο συμβαίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό φαλκιδεύει το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως γιατί είναι εκείνη η Ευρωπαϊκή Ένωση που επικρίνει το τι διαδραματίζεται σε τρίτες χώρες. Πρόεδρος. κύριος Φρουντσουλίτσα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας τον κύριο Παντσέρη γιατί πραγματικά ήταν τιτάνιο αυτό το έργο για την ετήσια έκθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και εκτιμώ ιδιαίτερο την η εισαγωγή του ε, για την πρόθεση των δικαιωμάτων των γυναικών, των παιδιών, των ε, θρησκευτικών, φιλετικών, εθνοτικών μειονοτήτων, γενικώ ε, τη πρόθεση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι μέλη μιας κοινωνίας παρόλο που υφίστανται εξαιρετικές ε, διακρίσεις ε, και στις περισσότερες χώρες χρήζουν ε, ιδιαίτερης κυβερνητικής προστασίας και υποστήριξη. Και εμείς θα πρέπει να γίνουμε υπόδειγμα με την προσέγγιση μας στο σώμα αυτό, γιατί οι κοινωνίες θα πρέπει να αλλάξουν από τη βάση και να γίνει σωστή διαπαιδαγώγηση για το σεβασμό των ελευθεριών. Επίσης, θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα παντού στην Ένωση, ώστε να μην χρειάζεται οι άνθρωποι να μεταναστεύσουν για να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά τους. Και επίσης, στη σχέση μα με τις τρίτες χώρες θα πρέπει να πετούμε πιο ε, αυστήρη τήρηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο συνάδελφος ο κ. Παντσέρη έκανε πολύ καλή δουλειά σε πολλά σημεία. Παρ' όλα αυτά έχουμε και κάποιες, ε, κάποιες επιφυλάξεις ε, διότι διαφωνούμε με ορισμένα πράγματα που λέει για τους πρόσφυγες, για την κλιματική αλλαγή, για το εξωτερικό εμπόριο και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία θίγει ο κ. Παντσέρη στην έκθεσή του. Η Λιθουανία, η Κροατία και η Σλοβακία ε, επικρίνονται για θέματα εσωτερικής πολιτικής. Πιστεύουμε ότι κάθε κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να αποφασίζει ε, περί των ε, οικογενειακών παραδόσεων στις οποίες θα μείνει προσιλωμένο. Υπάρχουν κράτη όπως στην Τουρκία που υποστηρίζουν το Ισλαμικό κράτος από την άλλη Κυρία Μπιλμπάου, Μπαραντέκα, Κυρία Μπιλμπάου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την γενοδορία σας. Η Ευρώπη θέλει να συνεχίσει να είναι σημείο αναφορά σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Για να το πετύχει, χρειάζεται μια ενιαία φωνή, και να είναι πιο γενναίες ό,τι αφορά της, ε, την προσήλωσή της. Ε, δεν είναι δυνατό να είμαστε δυνατοί και αυστηροί με τους πιο αδύναμους και μετά με τα πιο ισχυρά κράτη όπως οι ΗΠΑ, το Ισραήλ ή η Κίνα να είμαστε πιο χαλαροί. Αυτό εξηγεί και την χαλαρότητά μας σε ό,τι αφορά θέματα όπως η Παλαιστίνη ή η Δυτική Σαχάρα. Θα πρέπει άλλωστε να, τα του οίκου μας επίσης να είναι ξεκάθαρα. Γι' αυτό λόγο χρειαζόμαστε ένα σύστημα έγκαιρη προειδοποίησης όταν γίνονται σημαντικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. σήμερα είναι η Διεθνής Μέρα των Θυμάτων της Τρομοκρατίας και γι' αυτό λόγο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε την περικοπή των ελευθεριών ε, θα πρέπει όλη η Ευρώπη να στηρίξει τα θύματα της τρομοκρατίας μεταξύ αυτών και των θυμάτων τα οποία στην Ισπανία αυτή τη στιγμή έχουν αποτελέσει ήταν θύματα μιας, ε, ενός πραξικοπήματος και είναι θαμμένα σε τάφους που δεν γνωρίζουμε. Ο κύριος Χρυσόγωνος έχει το λόγο. Η απόψηνή μας συζήτηση είναι κάπως παράδοξη. Ασχολούμαστε με την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στον τρίτο κόσμο και δεν βλέπουμε τα προβλήματα μέσα στην ίδια την Ένωση. Στο βωμό της δημοσιονομικής σταθερότητας θυσιάζεται η δημοκρατική νομιμοποίηση αφού οι δυνατότητες καθορισμού πολιτικών από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια περιορίζονται ασφικτικά. θυσιάζονται όμως και τα θεμελιώδη ιδίως τα κοινωνικά δικαιώματα με τις διαρκείς περικοπές κοινωνικών δαπανών. εάν πραγματικά σας ενδιαφέρουν τα ανθρώπινα δικαιώματα θα σας συνιστούσα αντί να μακρηγορούμε για το τι συμβαίνει σε τρίτες χώρες να υλοποιήσουμε επιτέλους την προσχώρηση της ευρωπαϊκής ένωσης στην ευρωπαϊκή σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου και στον ευρωπαϊκό κοινωνικό χάρτη υποβάλλοντας έτσι τις πολιτικές της ένωσης στο διαρκή έλεγχο του ευρωπαϊκού δικαστηρίου δικαιωμάτων του ανθρώπου και της επιτροπής του ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη. τότε όμως οι ιέρακες της δημοσιονομικής πειθαρχίας εδώ μέσα θα δοκίμαζαν δυσάρεστες εκπλήξεις. Eh, eh, Κυρία Πρόεδρε, ε, το θέμα το οποίο συζητάμε είναι πάρα πολύ περίπλοκο και θα ήθελα να δείξω κάτι το οποίο δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα σε αυτή τη συζήτηση. Σε αυτή λοιπόν την έκθεση γίνεται αναφορά σε αντιτρομοκρατικές ε, δραστηριότητες. Και έχω την εντύπωση ότι όταν ε, αντιμετωπίζουμε τον, ε, την τρομοκρατία, η οποία μερικές φορές παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, κυρίως όταν πρόκειται για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας πω ότι εγώ δεν θέλω να θεσπιστεί ένα είδος πατριωτικής πράξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να αποφύγουμε να υπάρχει ένα είδος μεγάλου αδελφού και νομίζω ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε πιο στενά με το Συμβούλιο της Ευρώπης για να προετοιμάσουμε μια μακροχρόνια στρατηγική σε αυτόν τον τομέα. Πρόεδρος, ο κύριος Καστάλντο, τελευταίος ομιλητής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδης οι οποίοι εργάστηκαν για να υπάρξει αυτή η έκθεση που θεωρώ πράγματι ήταν πάρα πολύ κουραστική. Θα ήθελα να επενθυμίσω κάποια θέματα τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ. Θέματα όπου στο πρώτο σημείο γίνεται αναφορά στο ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας ε, νέος ε, κανονισμός ε, για τους ΛΟΑΤ και με βάση και το Διεθνές Δικαστήριο διότι κάποιοι οι υποψήφοι για να αποκτήσουν αυτό το κατεστώς. δεν πρόκειται για τη Σλόδα αλλά πρόκειται για τις υποψήφιους ε, τις, ε, που αναφέρονται στις γενικευμένες ε, πρωτεψηφιακές συμφωνίες. Εδώ επ' αυτού θα ήθελα να πω ότι όταν πρόκειται για ένα νομοσχέδιο νομίζω ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη αυτές οι γενικευμένες προτάσεις. Όλοι λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσαμε αυτό το θέμα να το αντιμετωπίσουμε με πολύ μεγάλη αυστηρότητα για τα κράτη-μέλη. Και το τελευταίο που θέλω να σας υπενθυμίσω είναι το 67, το άρθρο ε, έχουμε την γενοκτονία των Αρμενίων και σύντομα θα δοθεί ευκαιρία για να ε, εξοικειωθούν οι άμεσα εμπλεκόμενοι με το παρελθόν τους και να δουν και το τι μπορούν να κάνουν στο μέλλον. Πρόεδρος, ακούσαμε λοιπόν πολλές και λεπτομερές απόψεις και θα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Μοργκερίνη. Θα είμαι σύντομη, η συζήτηση ήταν ε, πολύ πλούσια, γεμάτη από σχόλια, προτάσεις, ε, υποδείξεις τις οποίες σημείωσα. Σας βεβαιώνω ότι ε, θα τις λάβουμε υπόψη μας ε, στην προετοιμασία των πολιτικών μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία τα, για τα επόμενα πέντε χρόνια. Θέλω να σχολιάσω ένα από τα πράγματα τα οποία, στα οποία αναφερθήκαν, αναφερθήκαν πολλοί από εσά. Δεν είναι κάτι το οποίο το συμπέραβα στις αρχικές μου παρατηρήσεις ε, και έχω ισχυρή προσωπική άποψη σε ό,τι αφορά τον ρόλο των γυναικών στην κοινωνία ε, σε ηγετικέ θέσει και σε ό,τι αφορά τη βία εναντίον των γυναικών. Είναι οι δύο πλευρέ του ίδιου νομίσματο. Οι δύο όψει του ίδιου νομίσματο. Ε, συμφωνώ με αυτό που είπατε ότι η καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών δεν είναι μόνο θέμα αλλαγής νομοθεσίας αλλά και σε μεγάλο βαθμό αλλαγής κουλτούρας. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε ε, από την παιδεία και όχι μόνο την εκπαίδευση των κοριτσιών, αλλά κυρίω την εκπαίδευση των αγοριών και στο σχολείο και στην οικογένειά του. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και στην εξωτερική μα πολιτική, αλλά και στι εσωτερικέ μα πολιτικέ. Ε, ε, αφιέρωσα τις εργασίε μας στις 8 Μαρτίου στι γυναίκε της, ε, του Αφγανιστάν και στα κορίτσια του Αφγανιστάν που ε, προσπαθούν να αποκτήσουν εμπειρία σε ηγετικέ θέσει στα θεσμικά όργανα, στην αστυνομία, ε, στο δικαστικό σύστημα, στα μέσα μαζική ενημέρωση. Θα πρέπει να τι υποστηρίξουμε και είναι πολύ ε, σημαντικό που τις καλέσαμε στα ευρωπαϊκά όργανα για ένα χρονικό διάστημα έτσι ώστε να μείνει ανοιχτό αυτό το κανάλι. Στις 9 Μαρτίου, την περασμένη Δευτέρα, δηλαδή βρέθηκα στη Νέα Υόρκη στις 8 Μαρτίου ε, συναντήθηκα με την ε, εκτελεστική για θέματα γυναικών του ΟΗΕ και συζητήσαμε το θέμα των γυναικών στις κοινωνίες, στην κοινωνία και το θέμα της βίας εναντίον των γυναικών μαζί με τον ε, Ευρωπαϊκό Ενταλμένο Ευρωπαίο ε, ε, ήμασταν παρόντες στην ε, CSW. Ε, θέλω να υπογραμμίσω λοιπόν τις πολύ χρήσιμες παρατηρήσεις σας. Ε, η δουλειά από τον συγητή είναι πολύ καλή και να αναλάβω δύο δεσμεύσεις και να σας δώσω δύο υποσχέσεις. Θα συντονίσουμε την δουλειά που γίνεται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεύτερον θα προσπαθήσουμε να επεκτείνουμε αυτή μας τη δράση σε όλους τους ε, τομείς. Ιδιαίτερος όταν εργαζόμαστε με τρίτες ε, χώρες σε όλο τον κόσμο και με τρίτους ε, θεσμούς. Ε, έχουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαφορετικά θεσμικά όργανα, αλλά η Κομισιόν θέλει να συνεργαστεί ιδιαίτερα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερα για τη συνεισφορά σας στη συζήτηση. Να ευχαριστήσω τους κοιόδης ηγητές και τον εισηγητή, τον κ. Πεντσάρη. Η έκθεση του αυτή είναι πολύ καλή. Θα αποτελέσει τη βάση για τις μελλοντικές μας εργασίε σε, αυτές τις, σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε. Ευχαριστούμε κυρία Ήπατη εκπρόσωπε. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο και στον εισηγητή μας τον κύριο Παντζέρη. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ λοιπόν όλους για τη συζήτηση και σας συγχαίρω για την ανανέωση της θητείας σας και συγχαίρω και σας κυρία Υπατή εκπρόσωπε γιατί θεωρώ ότι καταλάβατε τι είναι απαραίτητο να γίνει. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρχει μια διαφορετική ευαισθησία και θεωρώ ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι στο προήμιο του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων εκεί για άλλη μια φορά γίνεται λόγος για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο άτομο και επειδή μιλάμε για το άτομο εδώ δεν πρέπει να κάνουμε αφαίρεση αλλά ακριβώ το αντίθετο. Με τη λέξη άτομο θέλουμε να απομακρυνθούμε από αφαιρέσει ε, που είναι ε, το υποκείμενο ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να επισημάνουμε ε, το απαραβίαστο των δικαιωμάτων των όλων μας. Έτσι λοιπόν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπα, που άκουσα από τον Σοπράν Ντεμπράι, δηλαδή ότι είναι ε, ντροπή αυτά που ελέγχθησαν για τους ΛΟΑΔ και ε, μόνο σε επίπεδο ε, κοινωνίας των πολιτών νομίζω ότι μπορούμε να δείξουμε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Δεν είναι δυνατόν να πιστεύει κανείς το αντίθετο γιατί το αντίθετο σημαίνει ότι υπάρχει μυσαλλοδοξία. Έτσι λοιπόν απευθύνομαι στην ΚΟΥΑ, στην κυρία Βερζιά η οποία θεωρώ ότι θα πρέπει να σκεφτεί λιγάκι το θέμα της αποχής από την έκθεση παρότι τη σέβομαι. Θα ήταν παράδοξο με τον τρόπο αυτό να θέλει κανείς ε, να διαδώσει το σκοταδισμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό θεωρώ ότι η δουλειά που έχει γίνει είναι πάρα πολύ σημαντική και θεωρώ ότι η δουλειά αυτή θα τύχει της ε, μεγάλης ε, σύμφωνης γνώμης των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόεδρος, σας ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις ε, πληροφορίες. Έτσι λοιπόν έκλεισε τώρα αυτή η συζήτηση και τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα που επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό αλλά και δύσκολο παράλληλα θέμα και πρόκειται για την πολιτική ασφάλειας πιο συγκεκριμένα Πρόκειται για την αστατή κατάσταση στη Λιβύη και για τις συνέπειες